Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε συνάδελφοι. Και ευχαριστώ πολύ την συμπρόεδρο, την κυρία Κρέτσλε. Συνάδελφοι, όπως έτσι και αλλιώς ξέρετε, πρόκειται για μία συνέχεια της διερευνητικής έρευνας της Μαρτίνα Κουσναρόβα δημοσιογράφου. Έξι μέλη συμμετείχαν για την διερεύνηση αυτή. Ήταν εξαιρετικά σημαντική η αποστολή μας και γι' αυτό και είμαστε σήμερα εδώ. Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους των κρατικών αρχών, τοπικές αρχές, περιφερειακές, κοιό, δημοσιογράφους, ακτιβιστές και άτομα που διαμαρτύρονται Ιδιαίτερα εξετάσαμε θέματα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαίου και θα είμαι πάρα πολύ σύντομο γιατί ξέρω θέλω να μιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Καταρχήν, πολλοί ομιλητέ μας είπαν ότι υπάρχει δυσπιστία όσον αφορά του θεσμού και μεγάλη ανισορροπία μεταξύ της πραγματικότητας αλλά και των προβλημάτων που αφορούν ε, το κοινωτικό κεκτημένο. Βεβαίως το θέμα της προσφυγής στην δικαιοσύνη, οι δυσκολίες και τα προβλήματα όσον αφορά την ε, ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών, της καταπολέμησης της ε, διαφθοράς, της ανεξαρτησίας, των διερευνήσεων, συμμετοχή μαφίας, οργανωμένου εγκλήματος και οργανωμένου εγκλήματος στις συγκεκριμένες διαδικασίες. Όλα αυτά αναφέρθηκαν στην υπόθεση αυτή και βεβαίως ε, αυτό είναι κάτι που έχει ξεκινήσει και διερευνάται στην Σλοβακία και από διεθνείς υπηρεσίες πληροφοριών. Κυρία Γκρέσλε, πιστεύω ότι όσον αφορά τις ιδιαίτερες αρμοδιότητες της αποστολής αυτής, νομίζω ότι εσείς θα δώσετε περισσότερα στοιχεία. Αυτά είναι όμως σε γενικές γραμμές οι ανησυχίες μας και δίνω το λόγο στην Συμπρόεδρο. Ευχαριστώ. Από Σκοπιά Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού λάβαμε πάρα πολλές κατηγορίες από την ε, κοινωνία των πολιτών, βάσει των οποίων δεν παρακολουθούμε ε, υποθέσεις διαφοράς, σύμφωνα με τις απόψεις δηλαδή που εκφράστηκαν. Ε, αντιμετωπίσαμε και διάφορες φήμες σχετικά με την διασύνδεση της Ιταλικής μαφίας με την ε, Σλοβακία. Ασχοληθήκαμε και με το ερώτημα τι μπορεί να ήξερε αυτός ο δημοσιογράφος, τι μπορεί να ε, να διαπίστωσε κάτι, και τι μπορεί να ήταν αυτό που του κόστισε τελικά τη ζωή. Ε, συνδέεται κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι φαίνεται το θέμα με τα γεωργικά ταμεία και με την ε, διασύνδεση ε, της Σλοβακίας με την ε, Ιταλική μαφία. Τα διερευνήσαμε αυτά, συνεχίζουμε βεβαίως τη διερεύνηση αυτή της υπόθεσης. Είναι εδώ και μαζί μας εκπρόσωποι της Κομισιόν. Είναι χαρακτηριστικό το ότι υπάρχει, υπάρχουν μεγάλες ακαλλιέργειες ακτάσης στην ε, Σλοβακία. Ίσως και αυτό παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον. Υπάρχουν παρατυπίες στη Σλοβακία. Αυτό είναι γεγονός, αλλά ήταν γνωστές. Και από αυτή την άποψη η δική μας συνεργασία με τις λοβακικές αρχές ήταν καλή, αποτελεσματική και δεν υπήρχε λόγος ε, έλλειψης εμπιστοσύνη. Όμως ε, έχουμε ασχοληθεί και με το θέμα της ε, ανάπτυξης υπαίθρου. Πολλές φορές είχαμε γίνει παραλήπτες παραπώνων, σχετικά με παρατυπίες στις άμεσες ενισχύσεις και στα γεωργικά ταμεία γενικότερα στην Σλοβακία στις ε, άμεσες ενισχύσεις το ποσοστό σφάλματος είναι λίγο πάνω από το 2% στη Σλοβακία, λίγο πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, ε, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χωρίς όμως να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία που θα έπρεπε, κανονικά, που θα έπρεπε να μας είχαν οδηγήσει σε λεπτομερέστερη διερεύνηση ε, της υπόθεσης αυτής. Όπως και να έχει, η αποστολή αυτή ήταν πολύ σημαντική και νομίζω ότι η Σλοβακία θα συνεχίσει για πάρα πολύ καιρό ακόμη να μας απασχολεί. Ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διερεύνηση της Όλαφ για την Σλοβακία. Ε, κάτι που επίση είναι και αυτό στοιχείο ότι δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα γενικά στη χώρα. Πολλοί συνάδελφοι ε, είμαι βέβαιοι ότι θα θελήσουν να λάβουν το λόγο και γι' αυτό είναι σημαντικό ε, να τους δώσουμε γρήγορα το λόγο. Πρωτού δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους της Κομισιόν, θα ήθελα να ζητήσω από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας να μας πει ποια είναι η άποψή της για τα γεωργικά ταμεία και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στις άμεσες ενισχύσεις στην Ήπεθρο, ποια είναι τα προβλήματα οι ελλείψει, οι παρατυπίε που διαπιστώνονται. Περιμένουμε. Λοιπόν, η συνάδελφος Μέτσολα ζήτησε πρώτο το λόγο, επομένω ε, τον έχει. Παρακαλώ, κύριε Μέτσολα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω το λόγο για το επόμενο και όχι για αυτό και όχι αυτό το, σε αυτή τη φάση. Ναι, νομίζω είναι πολλοί συνάδελφοι που θα ζητήσουν το λόγο, οπότε να ολοκληρώσουμε τις αγωγικές μας παρατηρήσεις τώρα. Ολοκληρώθηκαν. Θέλετε να ξεκινήσει η Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Okay. So let's, let's go... Όχι, ας ακούσουμε πρώτα τους βουλευτές. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τους βουλευτές. Λοιπόν, η κυρία Μετσόλη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη. Νομίζω ότι θέλουμε να αποστείλουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ότι το Κοινοβούλιο πάντοτε θα διεκδικεί ελευθερία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προστασία των δεσιμογράφων. Όταν θανατώνεται ένας δημοσιογράφος, αυτό το είδους η εκτέλεση υπονομεύει τη δημοκρατία παντού. Και αν το επιτρέπουμε και δεν αλλάζει τίποτα στο status quo, και άλλα κρατημέλη θα ε, ρηπανθούν από το ίδιο τοξικό απόβλητο που ακολουθεί αναγκαστικά. Το μήνυμά μου εδώ λοιπόν είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά, να συνεχίσουμε να πιέζουμε ώστε τα κράτη-μέλη και οι πρόσωποι τους και κυβερνήσει κυβερνήσεις τους να κάνουν αυτό που οφείλουν. Ξέρουμε ότι πριν από έξι μήνες η Δάφνη Καρουάνα Γκαλίτσια δολοφονήθηκε στη Μάλτα γιατί έκανε αυτό που έκανε και ο Γιάνν Κουτσέκ στη Σλοβακία. Δηλαδή ε, αποκάλυπτε τις διασυνδέσεις μεταξύ βρώμικου χρήματος, βρώμικων τραπεζών και διεφθαρμένων πολιτικών, τα διαπλεκόμενα δηλαδή. Όλοι μας στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είμαστε εξαιρετικά πρόθυμοι να προστατεύσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι ε, αποφασιστικά για την ίδια την ύπαρξη της δημοκρατίας. Οι θεματοφύλακές τους έχουν απειληθεί και σε άλλα μέρη του κόσμου. Έχουμε εξεγερθεί κατά των ε, καταστολών αυτών επανειλημμένος εδώ για άλλα μέρη του κόσμου και οι ψευδείς ειδήσει καθώς και η παραπλάνηση στο ίντερνετ των ειδήσεων είναι στοιχεία που πρέπει να καταπολεμήσουμε εκεί όμως ιδιαίτερος όπου οι αρχές των κρατών μελών δεν κάνουν αρκετά για να αποκαλύψουν τους ε, εγκληματίες και την παράνομη δράση τους. Ευχαριστούμε κυρία Μπένοβα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για την οργάνωση της αποστολής στη Σλοβακία και όλος ιδιαίτερους τους συναδέλφους για την πολύ επαγγελματική τους συμπεριφορά. Ε, είχαμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε πολλές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής και θα ήθελα να σας ενημερώσω και για το τι αλλαγές έχουν προκύψει στη Σλοβακία από τότε που πήγαμε αυτή την επίσκεψη. Να σας πω τι έχει συμβεί λοιπόν. Στις 12 Μαρτίου ο Υπουργός Εσωτερικών ο Ρόμπερτ Καλνιακ, παρετήθηκε και στις 14 τρέχοντος παρετήθηκε και ο Πρωθυπουργός Φίτσο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε τον Πέτρε Πελεγκρίνη ως νέο πρωθυπουργό και ο Τόμας Τρούκερ έγινε υπουργό Εσωτερικών. Ακολούθησαν και άλλες αλλαγές και έχω αποστείλει μια ανακεφαλής αυτών των αλλαγών στη Γραμματεία. Ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για το τι συζήτησα σήμερα μόλις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών. προτάθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών ένα νομοσχέδιο που θα περάσει από τη Βουλή για να τροποποιηθούν οι διαδικασίες για τον διορισμό του αρχηγού της αστυνομίας, του επικεφαλής της αστυνομικής, των αστυνομικών δυνάμεων της χώρας. Κυρίως ε, για, την, ε, για τον αρχιεπιθεωρητή, τη θέση αυτή η εισαγγελία θα συνεργαστεί με την Ευρωπόλ και την ε, οργάνωση κατά της μαφίας της Ιταλίας ώστε να κάνουν μια κοινή έρευνα και να βρουν τη λύση σε αυτό το τραγικό ατύχημα στη Σλοβακία. Ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός μας πρέπει να λάβουν εμπιστοσύνη και αν η κυβέρνηση τους τη δώσει θα έρθουν σε συνάντηση με τους ευρωβουλευτές. Η αλλαγή αυτή έχει να κάνει ε, και με την ε, υπεξαίρεση κάποιων κονδυλίων που προορίζονταν για γεωργικούς σκοπούς. Ε, θα υπάρξουν λοιπόν ε, έρευνες και για το πώς έχει σχεδιαστεί η γεωργική πολιτική, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει καμία κατάχρηση των ε, κοντιλίων. Η Σλοβακία είναι η μόνη χώρα όπου υπάρχουν υποψίες για παράνομη χρήση κοντιλίων. Ήθελα λοιπόν να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς, την, προς τις οικογένειες του νεωρού αυτού δημοσιογράφου και της νηστής του, και να ευχαριστήσω τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, για την διοργάνωση αυτής της αποστολής και την όλη του εμπλοκή. Πρέπει η όλη υπόθεση να επιληθεί, αλλά πρέπει να επιληθούν και τα τρία ζητήματα που προέκυψαν σε σχέση με τις υποψίες για τη χρήση των κονδυλίων. Η νέα κυβέρνηση δήλωσε ότι υποστηρίζει όλες τις δράσεις ε, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αξίες της, οι οποίες θα ενσαρκωθούν και θα, ε, προσωπ... θα προωθηθούν από τη νέα ε, κυβέρνηση της χώρας. Ευχαριστούμε. Κύριος Γιάβορ, ευχαριστώ πολύ ως ε, συμμετέχον σε αυτή την επίσκεψη στην Σλοβακία. Πρέπει να πω ότι το σημαντικότερο για μας είναι να υπάρξει μια σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης ε, όσον αφορά τις ε, κατηγορίες αλλά και τα ανοιχτά ερωτήματα που συνδέονται με αυτό το τραγική ε, υπόθεση του δημοσιογράφου Κιούτσινια και της μνηστής του. Προφανώς επικεφαλής αυτών των ερευνών πρέπει να τεθούν οι, οι σλοβακικές αρχές χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ε, παρακολουθήσουν από κοντά την ε, εξέλιξη αυτής της έρευνας και βεβαίως να εξαρθούν και κάποια ευρωπαϊκά συμπεράσματα. Πρώτα, πρώτα απ' όλα πρόκειται για ένα περιστατικό που δεν είναι και το μοναδικό, σε μικρό χρονικό διάστημα μάλιστα, πρέπει να μας, ε, να μας κάνει να επικεντρωθούμε στην, ελευθεροτυπία, την ε, αποκαλυπτική δημοσιογραφία και το περιθώριο εντός του οποίου καλούνται οι δημοσιογράφοι να ε, εκτελέσουν το λειτουργήμά τους. Πρέπει λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να βελτιώσουμε την προστασία των αποκαλυπτικών δημοσιογράφων συμπεριλαμβανομένων κανόνων πανευρωπαϊκών σχετικών και να εγκριθούν οι κανόνες αυτοί το συντομότερο δυνατό προκειμένου να βελτιωθεί ε, η προστασία των δημοσιογράφων κάτι που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ως έργο από την πλευρά της Κομισιόν αλλά πρέπει να επιταχυνθεί. Επίσης πρέπει να ε, συσταθεί ένα χρηματοδοτικό μέσο για τα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την αποκαλυπτική δημοσιογραφία, κάτι που συζητείται ε, ζωηρά και εντό της Κομισιόν. Επίση, η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να ε, συστήσει βραβείο αποκαλυπτική δημοσιογραφία και νομίζω ότι και αυτό πρέπει να προχωρήσει. Το δεύτερο ζήτημα που επίσης είναι σημαντικό συνδέεται με το ζήτημα της διαφθοράς και εδώ πιστεύω ε, ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση στις σλοβακικές αρχές προκειμένου να προχωρήσουν στην, ε, σε βάθος διερεύνηση κατηγοριών που συνδύονται με πιθανή κατάχρηση γεωργικών κονδυλίων στην χώρα αυτή. Βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική έρευνα και του Όλαφ, είναι σημαντικό αυτό και με μεγάλη χαρά ε, θα δω και θα προτείνω και εγώ στην Επιτροπή να ζητήσει από το ελεγκτικό συνέδριο να προβεί σε έλεγχο των γεωργικών ε, ε, πληρωμών που έχουν γίνει στην ε, Σλοβακία σε ευρύτερο πλαίσιο και όχι μόνο στο πλαίσιο της συγκεκριμένη ε, υπόθεσης και να σκανάρουν όλες τις πληρωμές που έχουν γίνει στον, στη γεωργία, στον τομέα της γεωργίας στην Σλοβακία και επίσης πρέπει να ελέγξουμε αν οι μηχανισμοί σε ενωσιακό επίπεδο είναι επαρκείς για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της κατάχρησης των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όπως αυτό που φαίνεται να έγινε στην Σλοβακία, χωρίς φυσικά να είναι καθόλου η μόνη χώρα που πλήττεται από τέτοιου είδους προβλήματα ε, που συνδέονται με την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και τέλος, κάτι που θέλω και να προτείνω είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά να λάβουμε περαιτέρω πληροφορίες από τις ευρωπαϊκές και σλοβαϊκές αρχές και θα ήθελα να προτείνω να υπάρξει μια δεύτερη επίσκεψη των επιτροπών μας Λίμπε και Κοντ αργότερα εντός του 2018 προκειμένου να παρακολουθήσουμε και να σημειώσουμε την πρόοδο που θα έχει ε, πραγματοποιηθεί στην ε, Σλοβακία σε σχέση με την προηγούμενη επίσκεψή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκόμες. Σας παρακαλώ πολύ συνάδελφοι, σύντομα γιατί είναι και η Επιτροπή. Εγώ δεν ήθελα ε, να ενσωματώσω, δεν ενσωμάτωσα μάλλον, δεν συμμετείχα σε αυτή την αποστολή. Με ενδιαφέρει όμως ιδιαίτερα το θέμα. Υπάρχουν ε, νεκροί σε αυτή την υπόθεση και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία με αυτό που συνέβη στη Μάλτα με τη δολοφονία του δημοσιογράφου. Και πιστεύω ότι πραγματικά η παρακολούθηση του θέματος αυτού δεν μπορεί παρά να είναι ένα θέμα προτεραιότητας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πιστεύω ότι οι δύο αυτές αποστολές θα πρέπει κάπως να συνδυαστούν. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ανεξάρτητη και αμερόληπτη διαδικασία διερεύνησης. Πρέπει να πιέσουμε τις αρχές, γιατί αφού μας ζήτησαν τη στήριξη της Europol, και αυτό και στις δύο υποθέσεις, και στη Μάλτα και στη Σλοβακία, η Europol δεν θα πρέπει απλώς να συνοδεύει την έρευνα, αλλά να είναι ηγετικό ο ρόλος της στην διερεύνηση των υποθέσεων αυτών. Και εδώ δεν αναφέρομαι μόνο στην έρευνα για τη δολοφονία των δημοσιογράφων αυτών, αλλά και για την υπόθεση των Panama Paper. Η περίπτωση, αν θέλετε, της Δάφνη είναι κάτι που άμεσα σχετίζεται με τη διερεύνηση της υπόθεσης Panama Paper. Είναι λοιπόν καθοριστικό το θέμα αυτό. Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Όταν έχουμε ένα τέτοιο πραγματικό πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά έχει αγνοήσει και αρνείται να δεχθεί το πραγματικό πρόβλημα. Τώρα έχουμε υποψίες για την χρήση, την κατάχρηση αγροτικών κονδυλίων. Αλλά και στην άλλη υπόθεση, στη Μάλτα, υπάρχει ήδη ένα Άλλο θέμα που αφορά, όπως ξέρετε, τον Επίτροπο Ντάλι, ο οποίος αναγκάστηκε να παρετηθεί. Υπήρχαν υπόνοιες ε, διαφθοράς. Η κυβέρνηση όμως τι έκανε. Ουσιαστικά τον προστάτευσε. Έγινε σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Η Επιτροπή δε, δεν κούνησε το δαχτυλάκι της. Η Επιτροπή πρέπει πραγματικά εδώ βάση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς να είναι πολύ πιο δραστήρια, πολύ πιο αποτελεσματική και στις δύο αυτές τις υποθέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να στοχεύετε στην υπόθεση της Σλοβακίας όταν παίρνετε το λόγο και νομίζω ότι ήδη η αίτηση έχει γίνει στη Europol για να υπάρξει συνδυασμός ε, στις δύο αυτές έρευνες. Έχουμε ήδη ζητήσει και το ίδιο έχουμε κάνει και στις ε, αρχές της Σλοβακίας. Έχουμε βάλει ακριβώ το ίδιο αίτημα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκρέσλε. Πριν δώσουμε το λόγο στον επικεφαλής ε, για τα θέματα και στην Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Μάργαρετ Μπέτσον. Είμαι από την Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Η Ειδική Διεύθυνση για τις ασφάλειες και τον έλεγχο της Χριστοκονδυλίων. Βεβαίως και Υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα όσον αφορά τη χρήση των αγροτικών οικοδομών. Όμως δεν βρήκα πληροφορίες που μπορεί να μας βοηθήσουν για τις υποθέσεις αυτές και το τι ακριβώς συνέβη. Όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές, ναι, εκεί μπορεί να υπάρχει θέμα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ιδιοκτησία γης. Δηλαδή υπήρξαν κάποιες πληρωμές ε, που ε, αποδόθηκαν σε άτομα οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες της εν λόγω γης. Πέραν αυτού δεν βρήκα ισχυρά και τεκμηριωμένα στοιχεία για τις πληρωμές και τη χρήση των αγροτικών κονδυλίων. Για το θέμα της Σλοβακίας και τις άμεσες πληρωμές δεν έχουμε βρει δυσκολίες ούτε όσον αφορά τη διαχείριση ούτε τον έλεγχο των κονδυλίων τα θέματα της ιδιοκτησίας γης, των τίτλων, δεν είναι, όπως ξέρετε, κριτήριο αιρεσιμότητας και αρκεί αυτός που κάνει την αίτηση για τέτοιου είδους άμεσες πληρωμές και αγροτικά κονδύλια να έχει δικαιώματα για την χρήση αυτής της συγκεκριμένης γης. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι ο ιδιοκτήτης. Αυτό, αν θέλετε, ε, είναι το μόνο κομμάτι για το οποίο έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι διεθνείς αρχές βεβαίως, διοκτικές αρχές, μπορούν να διερευνήσουν αν υπάρχει εδώ άλλου είδους κατάχρηση ή ε, άλλου είδους παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Η αύξηση των δικαιούχων για τις άμεσες πληρωμές πάνω από 100.000 ε, ευρώ το χρόνο, αυτοί δηλαδή που μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία, για τους οποίους διαθέτουμε συγκεκριμένες πληροφορίες. Μεταξύ του 2015 και του 2017 δεν έχουμε παρατηρήσει συγκεκριμένες ε, διακυμάνθεις. Μόνο 40 επιπλέον δικαιούχοι έχουν προσθεθεί στην κατηγορία αυτή των ε, κονδυλίων. για το 2017 μάλιστα, για τις ε, κατηγορίες αυτές τις οποίες ελέγχεται, ενδεχομένως μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν 400 λιγότεροι δικαιούχοι από ό,τι στο 2015. Βλέπουμε λοιπόν εδώ η σύγκριση των στοιχείων μεταξύ αυτών που μας έχει υποβάλει η Σλοβακία και των στοιχείων που διαθέτουμε φτάνουμε στα ίδια συμπεράσματα όπως και η ελεγκτική υπηρεσία της ε, Σλοβακίας. Και τα θέματα αυτά είναι πολύ παρόμοια με αυτά τα οποία εμφανίζονται και σε άλλα κράτη-μέλη. Δηλαδή, κάποια κριτήρια αιρεσιμότητας, κάποια κριτήρια επιλογής, ε, κατηγοριοποίησης που δεν τηρούνται ακριβώς η τήρηση της νομοθεσίας για τις προμήθειες, για τη συμμετοχή. Αν θέλετε, σε σχέση με άλλες χώρες, συγκρίνοντας δηλαδή τα στοιχεία που διαθέτουμε για τη Σλοβακία, σε σχέση με άλλες χώρες δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές και διακυμάνσεις. Δεν έχουμε τίποτα λοιπόν που να μας ε, οδηγεί σε συμπεράσματα ούτε διαφθοράς ούτε μη κανονικών πληρωμών. Είχαμε επαφές με τις αρχές της Σλοβακίας από τότε που ήρθαμε εδώ στην Επιτροπή σας και σας υποβάλαμε μια πρώτη παρουσίαση για το θέμα αυτό. Και βεβαίως ε, εμείς οι DJ δεν είναι αρμόδια για παρακολούθηση και διερεύνηση τέτοιων θεμάτων. Οι μόνοι που μπορούν να το κάνουν είναι Όλαφ. Είπατε ότι χρειάζεται περισσότερος έλεγχος, κύριε Κιάβο. Οι μηχανισμοί ελέγχου διαρωτηθήκατε αν είναι αρκετά αποτελεσματικοί. Κοιτάξτε, εμείς σαν συνυπεύθυνη αρχή νομοθετική τηρούμε τις ισχύουσες ρυθμίσεις, κανονισμούς και νομοθεσίες. Οι έλεγχοι διεκπεραιώνονται λοιπόν βάσει αυτών των κανονισμών και σε γενικές γραμμές ήδη ε, μας επικρίνουν για εξαιρετικά επαχθείς αυστηρούς ελέγχους. Αυτό είναι, αν θέλετε, το σύνθεση σχόλιο που ακούμε από μέρους των κρατών μελών. Οι ελέγχοι υπάρχουν, οι ελέγχοι γίνονται, απευθύνονται στους δικαιούχους Και βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει κάποιος τους νόμιμους τρόπους να παρεκκλίνει κανείς ή να αποφύγει κανείς ε, την εφαρμογή. 7 εκατομμύρια δικαιούχοι υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της κοινή αγροτικής πολιτικής και το ποσοστό αυτών που προσπαθούν να αποφύγουν, να παρεκκλίνουν είναι ένα ελάχιστα χαμηλό ποσοστό, πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ενισχύεται τον εφιάλτη μου. Γιατί το, το χειρότερο που μπορούμε να πάθουμε είναι να έχουμε ένα νομικό σύστημα όπου υπάρχουν εθνικά παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται κάποιοι επιτίδοι. Ε, φαίνεται ότι μάλλον εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η δουλειά μας από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστούμε παρόλα αυτά και Βεβαίω θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα γιατί υπάρχουν κάποιε διαστάσει που θέλουμε να τι διερευνήσουμε και να τι φωτίσουμε σε μεγαλύτερη, ε, με μεγαλύτερε λεπτομέρειε. Βεβαίω θα ήταν και πολύ χρήσιμο ε, να μας πει και η αστυνομία ποιος ήταν ο τομέας στον οποίο ε, δραστηριοποιούνταν ο συγκεκριμένο δημοσιογράφος. Άλλωστε είχε λάβει και πολλά έγγραφα, είχε ζητήσει και είχε λάβει πολλά έγγραφα από την κυβέρνηση, Οπότε και όλα αυτά είναι στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν την υπόθεση ακόμη περισσότερο. Να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη γενική Διεύθυνση δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Δεν θα έπαιρνα το λόγο. Δεν έχετε τίποτα να πείτε. Of course we start... Ναι, βεβαίω μελετήσαμε την σχετική έκθεση πολύ προσεκτικά και σα ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά το μόνο που πρέπει να επισημάνω τώρα είναι ότι η Γενική Διεύθυνση Justice και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου εδώ και χρόνια αναλύουν τις εξελίξεις στο σύστημα δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και το 2016 και 2017 Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προτείναμε δύο συγκεκριμένες συστάσεις από τις αναχώρα συστάσεις για βελτιώσει στο σύστημα δικαιοσύνη τη χώρα αυτή, οι οποίε εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο και επικαιροποιήθηκαν για το 2018 ξανά στη σχετική έκθεση αναχώρα. Τον Μάρτιο για την ε, Δημοκρατία της Σλοβακίας συγκεκριμένα, όπου το θέμα της αρνητικής ε, εικόνας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναλύεται και εντοπίζεται, οπότε αυτό στην έκθεση, ίσω να μην τονίζεται αρκετά, όπω και στι συνομιλίε σα με του ενδιαφερομένους, η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή μελετάει τι εξελίξει στον τομέα αυτό. Και στι συναντήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνη. μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι στις συνομιλίες που είχαμε, κοιτάξαμε τι γίνεται και με την επικοινωνία τους με το Συμβούλιο της Ευρώπης και η σχετική έκθεση δημοσιεύτηκε στα περί Φεβρουαρίου. και από την DG Home η κυρία Γκεράη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω η έκθεση αυτή δείχνει ότι υπάρχει ήδη κάποια όθηση στην εξερεύνηση της υπόθεσης αυτής, όπως είπε και ο συνάδελφος του Γενική Διεύθυνση Τζάστ και εμείς ως Γενική Διεύθυνση παρακολουθούμε την εξέλιξη της διαφθοράς στην Σλοβακία με την σχετική έκθεση για τα θέματα αυτά, όπως και εδώ μια πενταετία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ε, αυτού του είδους ο διάλογος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ενισχύει το λένε και περισσότερο. Κάθε χρόνο είχαμε συστηματικά επισκέψεις και συνομιλίες με τις ε, αρχές και όπως και εσείς εντοπίσατε υπάρχουν συστημικά προβλήματα για τα οποία Κάναμε κάποια σύντομη ανάλυση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, αλλά η έκθεση αυτή ε, έτσι κι αλλιώς οδηγεί στις ε, ανασύσταση, αναχώρα συγκεκριμένα συστάσεις, ε, Οπότε σίγουρα όλα τα θέματα καταπολέμησης της διαφθορά στη Σλοβακία και μας ενδιαφέρουν και τα προσέχουμε με ιδιαίτερη Φροντίδα. Ναι, προ του ε, εκπροσώπου τη Γενική Διεύθυνση Home και Just ε, είναι προφανή κάποια από τα σχόλιά σα, αλλά καλό ήταν ε, που έγιναν στα πλαίσια αυτή τη επίσκεψη, τη αντιπροσωπεία μα, η οποία οργανώθηκε πολύ, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να ε, διερευνήσουμε το τι γίνεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα σε πολλές χώρες, όχι μόνο στη Σλοβακία. Έχουμε ένα τέτοιο μηχανισμό και προσπαθήσαμε εδώ να κάνουμε κάτι ε, πιο περίπλοκο, να συμμετάσχουν τέσσερις κοινοβουλευτικέ επιτροπέ στην αντιπροσωπεία για να καλύψουμε το σκέλο των κατηγοριών ε, τη της διαφθοράς καθώς και το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Από τη σκοπιά των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι κάποια από τα στοιχεία που ανακαλύψαμε επί τόπου δεν είχαν ε, να κάνουν μόνο με το τι συμβαίνει στη Σλοβακία. Το λέω αυτό για την Γενική Διεύθυνση Justice. Τέτοιε κατηγορίε ή τέτοιε καταστάσει εντοπίσαμε και σε άλλε χώρε με τα αρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνη. Οπότε έγιναν κάποιε συναντήσει, διεξοδικέ θα τι έλεγα, και θα έλεγα ότι η αντιπροσωπεία μα ήταν πάρα πολύ ε, προσεκτική στι ερευνέ τη. Υπάρχουν πολλά στοιχεία και στην έκθεση. βεβαίω. Το θέμα είναι ότι κάποιες φορές από τις διοκτικές αρχές και το σύστημα δικαιοσύνη της χώρας, οι έρευνες που γίνονται είναι πολύ ευρείες. Υπάρχουν όμως θέματα ελευθερίας του τύπου. Κάποια θέματα σαν αυτό δεν είναι κάτι που αφορά ειδικό στη Σλοβακία, αλλά μα ενδιέφερε να βρούμε τι είναι αυτό που κάνει την Σλοβακία διαφορετική ω προ τι υπόλοιπε. Ο κύριο κύριος α πούμε, αναφέρει το θέμα τη ελευθερία των δημοσιογράφων. Στόχο τη έκθεσης αυτή είναι να φύγουμε από εδώ, να πάμε και να σκεφτούμε πού μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει κάτι επιπλέον ω προ τη θέμενη αξία ευρωπαϊκή. Για την ελευθερία τη δημοσιογραφία, εδώ νομίζουμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωση με μια ευρύτερη προστασία ίσω σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό με ιδιαίτερη προσοχή και ω προ τις διαδικασίες δικαιοσύνη, τις δικαιοσύνης, δηλαδή τις δίκε, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις υπόλοιπε ρυθμιστικέ ε, αρμοδιότητες που μπορεί να έχουμε, δηλαδή τι διαδικασίες αναχώρα, ε, αναλύοντας την, ε, την πρόοδο τη κάθε χώρα και το σύστημά τη, το σύστημα δικαιοσύνη τη. Υπάρχει και αρμόδιος οργανισμός για αυτό και υπάρχουν και πολλοί τρόποι για να γίνει. Ε, στη σημερινή μας λοιπόν συνεδρίαση ε, να πω ότι με κάθε Υπουργείο της χώρας, με τις διοκτικές αρχές, τις αστυνομικές αρχές είχαμε συναντήσεις ιδιαίτερα διεξοδικές, συζητήσεις ιδιαίτερα διεξοδικές και είναι λίγο δύσκολο στην σημερινή μόλι συνεδρία να τα παρουσιάσουμε όλα αυτά. Όπω είπε όμω ο κύριο Γιάβορ για το θέμα των δημοσιογράφων, είναι σημαντικό η αντιπροσωπεία αυτή να το αφήσει αυτό παρακαταθήκη. Δηλαδή, να καταλάβουμε ότι κάποια από τα ζητήματα αυτά δεν αφορούν αποκλειστικώ και μόνο τη Σλοβακία, ειδικά για του δημοσιογράφου, να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αλλά αυτό εναπόκειται στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Η ελευθερία των δημοσιογράφων είναι κάτι που να το δούμε προσεκτικά και αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη ξεκινήσει και θα φροντίσουμε να υπάρξει σχετική συνεργασία με τι υπόλοιπε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ που ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά. Έχουμε κάποια κοινά εργαλεία για το θέμα της διαφθοράς, ε, στα πλαίσια της έκθεσης κατά της διαφθοράς, το ανέφερε η κυρία Γκόμες και άλλοι. Οπότε αυτό που προτείνω στους αδέλφους σήμερα, επειδή είναι πολύ ευρύ το πεδίο που καλύπτεται από όλα τα θέματα αυτά, και τις εξελίξεις ε, στη χώρα μετά την επίσκεψή μας. Όπως είδατε, εμείς τη δουλειά μας την κάναμε. Το κάθε θέμα που μας ζητήθηκε το ε, θίξαμε. Σωστά λοιπόν ε, ανέλαβαν οι δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Τώρα οι υπόλοιπε που πρέπει θα εγκύψουν στα θέματα αυτά και για το θέμα των δημοσιογράφων θα δούμε κατά πόσον υπάρχει απέτηση να πάμε παραπέρα. Ως προς την πρακτική εφαρμογή να υπογραμμίσω ότι η αντιπροσωπεία δεν δίστασε να υποβάλει προτάσεις, συστάσεις σε κάθε ευκαιρία. Παρόλο λοιπόν που υπάρχει διεθνή συνεργασία για τη συγκεκριμένη έρευνα, εμείς αμέσως ζητήσαμε κοινή ομάδα έρευνας. Γιατί θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν προς όφελος και της ίδιας της Σλοβακίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, νομίζω ότι λοιπόν τη δική μας προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία την προσφέραμε στη χώρα. Ε, και η αντιπροσωπεία μας έκανε ό,τι μπορούσε για Ε, το έχω πει και σε προηγούμενες ε, συναντήσεις. Η χώρα βρισκόταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση αυτές τις μέρες. Τα μαθήματα που πρέπει να αντλήσουμε από όλη αυτή την εμπειρία είναι διαφορετικά για κάθε επιτροπή αλλά να το πω γιατί ήταν εδώ η Γενική Διεύθυνση Home και Just με μία δήλωσή τους. Σίγουρα τα θέματα αυτά ειδικά πως αλλά πρέπει να του δώσουμε και μια ιδιαίτερη φώτιση αυτή τη στιγμή με αυτά που έχουν συμβεί. Αυτό είναι το σημαντικό για την Επιτροπή Λίμπερ. Ευχαριστώ. Έτσι και αλλιώς η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα παρακολουθήσει την ε, ήδη συγκεκριμένη διαδικασία όπως έχει ξεκινήσει. Ο Μάρτιος είναι ένας δύσκολος μήνας, έχει σχεδόν τελειώσει έτσι και αλλιώ. Είμαστε σχεδόν στον Απρίλιο και βεβαίως ε, θέλουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τις ανάγκες αυτής της χώρας, η οποία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε περισσότερη ασφάλεια, συνείδηση και θα πρέπει ο Ευρωπαίος Φορολογούμενος να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει με τα χρήματα του και βεβαίως ε, αυτές οι δολοφονίες ε, θα πρέπει να διαλευκανθούν γιατί έχουν άμεση σχέση και με αυτό. Είναι 6.30, μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μας. Σας εύχομαι σε όλους καλό βράδυ.